Διαδικαστικό η κυρία Ζούμπερ. Κυρία Πρόεδρε, θα ψηφίσουμε τρία ψηφίσματα από τα κατεπήγοντα και θα τα ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς με ονομαστική ψηφοφορία που θα καταχωριστεί. Διεκδικούμε το δικαίωμα να μπορούμε να κάνουμε και γραπτές δηλώσεις και να εξηγήσουμε γιατί ψηφίσαμε έτσι αλλιώς. Αυτό το θεωρούμε παράδεκτο. Θα πρέπει αμέσως να αλλάξουν οι κανόνες, ώστε να μπορεί ένας βουλευτής να κάνει την επεξήγηση ψήφου για τα θέματα αυτά όπως προβλέπετε. Η Πρόεδρος.